Uh, uh, Κυρίες και κύριοι, καθίστε παρακαλώ για να αρχίσουμε την ψηφοφορία. Το πρώτο θέμα που θα ψηφίσουμε είναι το ψήφισμα σχετικά με τη σύλληψη του Αλεξέη Ναβάλνη και άλλων διαδηλωτών. Από ό,τι καταλαβαίνω θα υπάρξει ψήφισμα βάσει του άρθρου 194 και θα δώσω το λόγο στον κύριο Σόλτς. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι.